αφορά τώρα τον ορισμό εισηγητών και συντακτών γνωμοτοδοτήσεων. Έχουμε την σύσταση των συντονιστών ε, για την οδηγία καταρχήν η οποία τροποποιεί το ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης των ναυτικών πάει στον πρόεδρο όπως επίσης και η επόμενη έκθεση όσον αφορά τα πετρελοφόρα Καδίκοκα γιατί καμία ομάδα δεν εξέφρασε ενδιαφέρον, οπότε τα αναλαμβάνει ο πρόεδρος. Έρχομαι τώρα στις γνωμοδοτήσεις. Οι γνωμοδοτήσεις θα γίνουν ως εξή εξαιτίας του συστήματος περιτροπής που έχουμε. Αλλά υπενθυμίζω στους ευρωβουλευτές ότι οι γνωμοδοτήσεις αναφέρονται εδώ με την σειρά που τις παίρνουμε, για να είμαστε δίκαιοι. Οι γνωμοδοτήσεις έχουν ως εξή λοιπόν. Ε, σκάφη αναψυχής, το ECR. Η απαλλαγή 2010 του Γενικού Προϋπολογισμού το αναλαμβάνουν οι σοσιαλιστές. Έπειτα οι συντονιστές συμφώνησαν τα σημεία 5, 6, 7 και 8 που είναι απαλλαγές για τις διάφορες ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες να εξεταστούν σε μία γνωμοδότηση που αναλαμβάνουν οι σοσιαλιστές. Συμφωνήσαμε επίσης τα σημεία 9, 10 και 11 διαρθρωτικά ταμεία και ταμείο συνοχής επίσης να εξεταστούν σε μια γνωμοδότηση που αναλαμβάνουν οι πράσινοι. Για τα έγγραφα τώρα τα οποία φτάσαν σε εμά προς ενημέρωση πρώτα απ' όλα έχουμε την πολιτική πορεία με το Αζερβαϊτζάν και εδώ εκ περιτροπής αποφασίζεται το ποιο αναλαμβάνει συντάκτη. Οι πράσινοι λοιπόν αναλαμβάνουν το σημείο 12 και το σημείο 13 εδώ δεν θα κάνουμε τίποτα, έτσι αποφασίσαμε. The Οι συντονιστές επίσης πήραν και τις εκθέσεις όσον αφορά την επιτροπολογία. Συζητήσαμε τις διάφορες ιδέες για συνεργασία με άλλα κοινοβουλευτικά σώματα και καταλήξαμε σε ποιους τομείς θα θέλαμε ε, τέτοιες ε, σχέσεις με άλλα κοινοβουλευτικά σώματα. Και αυτό είναι το ρικάστη για τους σιδηροδρόμους. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Το πακέτο αεροδρομίων, ECR και τα βιώσιμα κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές για τη συγχρηματοδότηση των TEN-T. Η εφαρμογή επίσης όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών διασυνοριακά για όλες τις μορφές μεταφορών και η ανάπαυση των, φορτηγών, των οδηγών φορτηγών. Εδώ θέλουμε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα φροντίσουμε να γίνει αυτό στη βάση που έχει γίνει και κατά το παρελθόν, που είναι να χρησιμοποιούμε τους ε, συντάκτες μας, αυτοί οι συγητές μας δηλαδή, θα έρχονται σε επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουμε. Επόμενο θέμα τώρα ήταν έτοιμα που μας ήρθε Όσον αφορά τους ταχυγράφους, ζητήθηκε, προτάθηκε η κυρία Τικάου να έχουμε μία μήνυα κρόαση για αυτό το θέμα. 20-21 Δεκεμβρίου. Ταχυγράφη λοιπόν. Επίσης θέλω να σας πω αυτό που είπα και στους συντονιστές. Ότι δηλαδή πολλοί από εμά υποστηρίζουμε τι μήνυ ακρόασει, αλλά πολύ λίγοι από εμά είναι παρόντες στις ακρόασει. Αν αποφασίσουμε για ακρόαση, λοιπόν, σα παρακαλώ να είσαστε παρόντε. Οι συντονιστέ επίση αποφάσισαν ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πιο θετικό και επικοδομητικό όσον αφορά την εβδομάδα κινητικότητας του 2012. Συμφωνήσαμε επί της αρχής και θα προταθούν ιδέες στη συνέχεια. Στη συνέχεια θα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση συντονιστών στο Στρασβούργο στις 26 του μηνός για τα 10 όταν θα έχουμε επίσημα πάρει πια την πρόταση της Επιτροπής. Θα έχει συμφωνηθεί στις 19 του μηνός κανονικά από το Σώμα των Επιτρόπων. Και συμφωνήσαμε επίσης ότι πρέπει να ακολουθήσουμε να παρακολουθήσουμε την παρέμβαση για Ζεμπόφσκι και οι συντονιστές θα προτείνουν πράγματα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περισσότερο και για το ΦΑΠΑ και για το SES2 για να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς θα προχωρήσουν μετά την έγκριση. Αυτά είναι βασικά που έχω να σας πω όσον αφορά τη συνεδρίαση των συντονιστών. Κυρία Φώστερ, σας ακούμε. Όχι για την ε, συνάντηση αυτή, αλλά πρόεδρε, μια που θα ψηφίσουμε για πολλή ώρα. Δεν σας ακούω πολύ καλά χωρίς τα ακουστικά μου. Δεν με βολεύουν να τα φοράω, βλέπετε. Ε, μια που μπορώ να σας καταλάβω χωρίς ακουστικά, μήπως γίνεται να δυναμώσουμε λιγάκι την ένταση ώστε να μπορώ να σας ακούω χωρίς να χρειάζεται να φοράω τα ακουστικά μου. Πρόεδρος, εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάπως αλλιώς. Εγώ από εδώ δεν μπορώ να δυναμώσω τον ήχο. Ποτέ δεν με κατηγόρησε κανείς ότι δεν ακούει τη φωνή μου αρκετά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Θα προσπαθήσω πάντως να μιλάω πιο δυνατά, λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνείτε λοιπόν όλοι για το σας είπα, για τους συντονιστές, τις συστάσεις τους, εντάξει. Ωραία. Κύριε Κιμουτσάκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητάω το λόγο. Ξέρω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη και μακριά ψηφοφορία. Ζητάω το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου που εργάστηκαν, ειδικά του συντονιστέ, που εργάστηκαν με πνεύμα επικοδομητικό αλλά και με αποφασιστικότητα για να κλείσει το θέμα ε, ε, του κειμένου για την ενιαία θαλάσσια πολιτική. Ε, και πάλι ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κουμουτσάκο και για το έργο σας. Ωραία, συμφωνήσαμε με αυτά. Αλλάζω χαρτιά εδώ μπροστά μου. Και περνάμε στις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία που έχουμε είναι Α, το κάναμε αυτό κύριε Κουμτσάκο. Πήγα να πω το δικό σας θέμα, αλλά ήρεμα, ήρεμα. Δεν έχουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική τώρα, εντάξει, νόμιζα θα το ψηφίζαμε τώρα. Όχι, recast λοιπόν. Αναδιατύπωση, εντάξει. Συμφωνείτε όλοι. Πω, πω. Τι είσαστε εσείς. Σύμφωνοι. Να σας πω ότι οι τροπολογίες αναλαμβάνονται από τον κύριο Τιμπάκερ. Είναι 283 μέχρι 291. Εντάξει. Ας κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να ξέρουμε ότι δεν κλέβει κανείς. Μην είσαστε παραπάνω από όσοι θα έπρεπε. Για να ξεκινήσουμε αυτή τη δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε η ψηφοφορία. Πέρασε. Για, απαντέψτε ποιος, ποιοι έχουν ψηφίσει παραπάνω πώς θα έπρεπε. Το ΕΛΚ. Ματιέ, παραπάνω. Ένας. Εντάξει, ξεκαθαρίστηκε. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, εντάξει τώρα. Αρχίζουμε. Άρθρο 2. Πρώτη παράγραφος. Να είσαστε λίγο υπομονετικοί πάντως. Όπως ξέρετε είναι περίπλοκη η ψηφοφορία και μπορεί να χρειαστεί να συζητάμε εδώ στο στέδρανο αυτό για να συμφωνήσουμε ποιο είναι το επόμενο που πρέπει να ψηφίσουμε. Λοιπόν, θα σας λέω κάθε φορά τι ψηφίσουμε. Άρθρο 2, παράγραφος 1, τροπολογία 254 της κυρίας Βουίλς υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 255, υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 256 Will υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 261. Υπάρχει προφορική τροπολογία αριθμός 9, Μαρκίνκοβιτς και Ζασάντα. Αντιρρήσεις. Αν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροποποίηση, πείτε το. Ε. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι, ωραία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 261 με την προφορική τροποποίηση. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της προφορίας. 20 υπέρ, 23 κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα το 261 χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 263. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Χωρίς το κομμάτι που λέει σε ένα δίκτυο το οποίο κτλ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα με τις λέξεις αυτές υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 του συγκητή με προφορική τροποποίηση 1. Καμία... Όχι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. 267, ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 268 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 2, παράγραφος 4. Έχουμε μια προφορική τροπολογία αριθμός 2 του κ. Μαρουνέσκου. Έχετε καμία αντίρρηση? Παρακαλώ, ο κύριο Σέινταλ Καντραουή. Ναι, εμεί έχουμε αντίρρηση. Γιατί πηγαίνει υπερβολικά μακριά. Ωραία. Συνεπώ αφού υπάρχει αντίρρηση, δεν μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε. 269. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 272. Προφορική τροπολογία αριθμό 3 του εισηγητή. Αντιρρήσεις. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεπώς, συνεχίζουμε και φτάνουμε 274. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα είναι το 2α αριθμιστικό σώμα που σημαίνει κτλ. Και το δεύτερο τμήμα είναι και επίσης από το τμήμα πολιτικής. Λοιπόν, το πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο τμήμα της 274. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα που πρέπει να ψηφίσουμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. 275. Κύριε Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 276 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 278 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 279 κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Το πρώτο περιφερειακές υπηρεσίες και μετά διαγράφει αυτό που βλέπετε μπροστά σας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 280 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 282 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 284 κατά τμήματα ψηφοφορία. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα το βλέπετε υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 283 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 281 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ για το 285. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις προφορίες. Μεταξύ δύο γουλιών τσάι. Απορρίπτεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είμαι σίγουρος, ξανά, 290 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 293 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 295 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 296 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 297 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 298 και 299 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική α. Συμβιβαστική α εκτός τα δύο τμήματα που βλέπετε που αναφέρονται στα εισοδήματα άλλων συνδρομικών επιχειρήσεων. Υπέρ της α λοιπόν, της συμβαστικής α. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε τις δύο αυτές παραγράφους. Την πρώτη πρώτα για τα εισοδήματα των συνδρομικών επιχειρήσεων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και τώρα τη, η παράγραφος 4 με τις διατάξεις αυτές υπέρ, κατά, αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την παράγραφο αυτή 4, τελευταία πρόταση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη σελίδα 9. Συμβιβαστική τροπολογία Β. είναι υπέρ της συμβαστικής Β παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στις χωριστές ψηφοφορίες. Η τρία αποζητήθηκε από την ΚΟΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη δεύτερη χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ ψηφίζουμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία αριθμός 2 που ζήτησε η Άλντε ψηφίστε παρακαλώ Άλντε, Άλντε φιλελεύθερον χωριστή ψηφοφορία ρυθμός 2 για να εγκριθεί μία παράγραφος 3α νέα που λέει και ρήτρε ασφάλειας για τις υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τώρα έχουμε πάλι μια χωριστή ψηφοφορία από την ΚΟΕ για την αντιλογική σκέψη ΠΕΡ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στη σελίδα 11. Τροπολογία 291 που είναι τελευταία σε αυτή τη σελίδα του κύριου Στέρξ. 291 άρθρο 4 παράγραφος 2 β νέα. Διαφωνείτε κύριε Σιγητά. Μπορεί να είναι σε άλλη σελίδα, τι να πω. Σε μένα είναι σελίδα 11, είναι άρθρο 4, παράγραφος 2β9, τροπολογία 291 του κυρίου Στέρξ. Μας άφησε κληρονομιά, τι να κάνουμε. Σύμφωνοι, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές θα το ελέγξω, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ για το 291 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία Γ. Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 357 τώρα στη σελίδα 13 τουλάχιστον στο δικό μου κατάλογο, άρθρο 9, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2. Τικάου. Συμφωνεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 358. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 360. Έχει αποσυρθεί. Παράβαση εκτός μικροφώνου. Απορρίφθηκε. Α, 358 θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Ψηφίζουμε λοιπόν. 358. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίνεται. Αλλά δεν ήταν αυτό που δείξαν τα χέρια που σηκώθηκαν πριν. αλλά δίκαιο είχατε που ζητήσατε να ελέγξουμε. Αλλά σας επαναλαμβάνω δεν δείξαν αυτό τα χέρια. 359 τρεμόσα η βάλση με προφορική τροποποίηση 4 δεν υπάρχει αντίρρηση. Ωραία ψηφίζουμε λοιπόν. Α κύριε Κόλτσεκ έχετε αντίρρηση στην προφορική τροποποίηση. Εντάξει. Συνεπώς ψηφίζουμε την 359 χωρίς την προφορική τροποποίηση με το International μέσα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 361 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 362 έχει αποσυρθεί, 363 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 364 έχει αποσυρθεί, 365 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 366 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 367. 368 και 369 γιατί είναι ίδιες υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτονται 31 του συγκεκριμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 370 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα. 370, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της φοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 372. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 374. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 373. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 375. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 378 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ για την 378 Ψηφίστε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 379. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 385 και 384 που είναι ίδιες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 33 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 386 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 387 και αποσυρθεί. 388 με προφορική τροποποίηση 5 αντιρρήσεις για την προφορική αυτή τροποποίηση. Όχι. Ωραία. Με την αλλαγή αυτή υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε. Συμβαστική D. Με μία σειρά από χωριστές ψηφοφορίες που έχουν ζητηθεί και υπάρχει και προφορική τροπολογία 6, αντίρρηση, βλέπω τον κύριο Κόλτσεκ. Δεν μπορεί να γίνει ψηφοφορία στην προφορική τροποποίηση 6. Συμβιβαστική D χωρίς την προφορική τροπολογία ε, ψήφι κατά, απόχες. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία για την προφορική. Όπα, όπα, όχι για την προφορική 6, για τη συμβαστική D, λέει και πάλι ο πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Χωριστέ ψηφοφορία τώρα. Για την παράγραφο 2 και 4 η δεύτερη πρόταση από την ΚΟΕ ψήφισε κατά αποχές εγκρίνεται. 3 των πρασίνων στην παράγραφο 2 και παράγραφο 4 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία 4 για την ΚΟΕ Παραφώς 2 και παραφώς 4 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία για τη χωριστή ψηφοφορία υπαριθμών 4. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Χωριστή ψηφοφορία 5 γκουε. Παράφος 2 και υποπαράφος 5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία 6, γκουε, παραφος 3 και 4, ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε τώρα. Είναι σελίδα 22 στο δικό μου κατάλογο, ίσως είναι 23 στο δικό σας. Είναι σφιχτή η τυπογράφηση στην ομάδα του ΕΛΚ. Ή μάλλον πρέπει να γίνει πιο σφιχτή. Right. Because we have agreed the same wording in the... Επειδή έχουμε ήδη αποφασίσει μια διατύπωση στην προηγούμενη συμβαστική τροπολογία, δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε Όλε αυτέ τι χωριστέ ψηφοφορίε γιατί τι έχουμε περάσει ήδη. Ψηφίσουμε απλώ τη συμβαστική ε. Όλο το κείμενο, συμπούρμπουλο, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 456, σελίδα 25. Στο κείμενο του Πρόεδρου τουλάχιστον. 456 για το άρθρο 14 παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 457 υπέρ κατά αποχές μήπως μπορούμε να ελέγξουμε την 457 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίθηκε. 458 υπέρ κατά θα ξαναδοκιμάσω. Αρχίζει η χεροκούραση τώρα. Ψήφι υπέρ της 458. Κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λόγω κόπωσης βραχιώνων. Άρχεται η ψηφοφορία για την 458. Ψηφίσατε όλοι πέρα τη ψηφοφορίες. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 459 υπέρ. <clears throat> Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 του της ηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΦ. για το άρθρο 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 102 άρχεται. Πρόκειται για το παράτημα 4. Ψήφισατε όλοι ε, Πέρασε η Απορρίπτεται. 103 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 477 σελίδα 27 στο έγγραφο του Προέδρου 477 στη, στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 478 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 479 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 εισηγήτρια ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 480 τρώει χώμα τις υπόλοιπες μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινό από τη 49 ως την 104 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 482 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκπίπτει 483 πάμε στη 485 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 συγγήτριες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 486 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. 484 εκπίπτει. 487 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 συγκίτρες και 488 επταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε 56 και 48 από κοινού άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, όλες, πέρας. Απορρίφθηκαν. 57. <clears throat> Εισηγήτριας, υπέρ. Α, πήδηξα 489. 489. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57. Ψήφι υπέρ κατά έλεγχος για την 57 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται η 490 εκπίπτει 491 βαντάλεν ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από την 58, 105, 106, 107 λοιπά μέχρι την 111, όλες από κοινού ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. 693 και 6 εκπίπτουν, 492 υπέρ, ψήφι υπέρ και 43 κατά, απόχες απορρίπτονται. Και η 495 Αγιάλα Σέντερ, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτων. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 59 <clears throat> της εισηγητρίας υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G όπως το γκολφ. Ψήφι Κατά. Αποχές. Εν κρίνεται. Συμβιβαστική H. Στην 31 στο δικό μου κείμενο. Σελίδα 31. Και έχουμε κάποιες χωριστές ψηφοφορίες όπως ήθιστε. Πρώτα η προφορική, πρώτα και μια προφορική τροπολογία. Πρώτα η συμβαστική τροπολογία όπως έχει υπέρ κατά αποχές δεκτή. Χωριστή ψηφοφορία 1 της ΓΚΟΕ ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρόφορική τροποποίηση 7 των πρασίνων υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ψήφι υπέρ. Κατά. αποχέσενγκ. Μπορούμε να ελέγξουμε. <clears throat> Προφορική τροποποίηση 7 των πρασίνων. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 22-20. Χωριστή ψηφοφορία 2 από την ΚΟΕ. Παράγραφος 7, πρώτη παράγραφος, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε την χωριστή ψηφοφορία 2 της Γκουε άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρασε προκτηριες 37-7 εγκρίνεται αρχίστε να κουράζεστε βλέπω χωριστή ψηφοφορία 3 της Γκουε ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται χωριστή ψηφοφορία 4 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην συμβιβαστική I στη σελίδα 34. Το ΕΛΚ είναι δύο σελίδες μπροστά από ό,τι βλέπω. Συμβιβαστική I, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία. Των πρασίνων ένα, ψήφι υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερη χωριστή ψηφοφορία των πρασίνων στην παράγραφο 5 ψήφι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Πάμε στην 547. Στη σελίδα 36. Αυτό 35 παράγραφος 1. Κράμερ Ντουράν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού την ε, συμβαστική τροπολογία μαζί με τις τροπολογίες 68 και 123, 123, 124, 125 ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρέθησαν. 549 και 7-16 εκπίπτουν 5-48 κραμεντυρά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5-5-2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5-3 έχει αποσυρθεί 5-5-4 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 556 καθώς και 557 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε 556 και 557. Άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκαν στο τσακ. Οι 555 και 558 εκπίπτουν. Πάμε στην 559 για Λασέντερ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 561 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 562 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 563 και 564 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 70 της εισηγήτριας και 565 ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 567 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 568 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 569 και 570 είναι ταυτόσιμες. Ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 571 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 572 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 573 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 574 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 575 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 576 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 577 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 570 8 Φαντάλεν, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 <clears throat> της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 579 υπέρ κατά αποχές δεκτή 580 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 581 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 582 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 583 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 584 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική K ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Συμβιβαστική L στη σελίδα 40 του Πρόεδρου. Και έχουμε τέσσερις χωριστές ψηφοφορίες. Καταρχήν όμως κάνουμε τη συμβαστική L, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Χωριστή ψηφοφορία ένα γκουε. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Χωριστή ψηφοφορία της 1 της Γκουε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 39-4. Μάλιστα. Το ΕΛΚ δεν ψήφισε γι' αυτό. Χωριστή ψηφοφορία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Χωστή ψηφοφορία 3 της ΚΟΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Split vote 4 χωρίς ψηφοφορία 4 ΚΟΕ υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίνεται. Συμβιβαστική M Εντάξει, τη βρήκατε. Συμβαστική M, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική N τώρα. ψήφι υπέρ συμβαστικής N. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. τροπολογία 89 της κοινού αποκινουμε Αποκινούμε 90-91 μέχρι τη 2 μέχρι την 14 και τη 252. Μέχρι την 14, συγγνώμη, της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 252 εκπίπτει και η 643 εκπίπτει. 69 και 71 από κοινού, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Εκπίπτουν οι 550 και 551. Πάμε στην 566, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 644, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 94 έως 98 και 15 unblock ψήφι κατά αποχές εγκρίνονται 645 εκπίπτει 646 ψήφι κατά αποχές εγκρίνονται. 647 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική Ο. Με χωριστή ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Πρώτα συμβαστική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η χωριστή ψηφοφορία του ΕΛΚ για την Παύλα 11. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική π Τη βρήκατε για το παράδειγμα 7. Και εδώ υπάρχει χωριστή ψηφοφορία. Πρώτα συμβαστική τροπολογία ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία των φιλελευθέρων ψήφι υπέρ κατά αποχές. Μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Χωριστή ψηφοφορία των φιλελευθέρων της άλδε στο, στο παράτημα 7. Ψηφίσατε όλοι. πέρα της ψηφοφορίας. Περνάει. 34-9. Συμβιβαστική Q. Ονομαστική κλίση από τους πρασίνους έχει ζητηθεί, οπότε κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία ούτως ή άλλως. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Συμβαστική Q για το παράτημα 8.1. όνομα κύκλη σα πενθυμίζω. τον των πρασίνων. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία. τη ψηφοφορίας. 28-11 έχει εγκριθεί με μία αποχή. Συμβιβαστική R στο παράτημα 8-5 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 7-21, η Μπρασάς και το παράτημα 9 ψήφι υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 7-22, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 723 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 724 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στις αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Ξεκινάμε με την αιτιολογική σκέψη α, μικρό α, τροπολογία 130 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του συγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 141. Θα ελέγχουμε για την 140 του κυρίου Κράμερ. Τροπολογία 140. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 141 του κυρίου Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε για την 141. Όλο και λιγότεροι σηκώνουν τα χέρια τους. Ξέρω ότι κουράζεστε σιγά σιγά. Ελέγχουμε για την 141. Υπάρχει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 150 ηλεκτρονική επαλήθευση άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την τροπολογία 4 του εισηγητή άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε για την 155 άρχιτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 157. Με συγχωρείτε. Απορρίφθηκε με δύο ψήφους. 21-23. 21 υπέρ, 23 κατά. Είμαστε στην 157 τώρα, υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 157 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 19 κατά. 161 υπέρ. Μάλλον καταπίπτει, με συγχωρείτε, 161. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159 χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα, χωρίς την διατύπωση The Existing National, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν καταπίπτει. Έτσι, όχι, μάλλον πρέπει να ψηφίσουμε και το δεύτερο τμήμα, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε λοιπόν το δεύτερο τμήμα, These Words Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Έχει αποσυρθεί το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από τους πρασίνους για τις επόμενες τρεις τροπολογίες. Περνάμε στην 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 163 υπέρ κατά αποχές Α ελέγξουμε για την 163. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε. Άρτη ψωφορία, Πέρας. Και όντως απορρίπτεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, ας το επαληθεύσουμε. Πρέπει να σας πω όμως ότι τα τρία τέταρτα του ΕΛΚ δεν ψήφισαν. Αν λοιπόν δεν νοιάζουν να ψηφίσουν, τι να σας πω, επαληθεύουμε πάντως για την 165. Πάντως διανατάσεως το αποτέλεσμα ήταν σαφές. Άρτη ψηφοφορία για, για την 165. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 327 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 166, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 170 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι επόμενες, οι επόμενες δύο καταπίπτουν. Πάμε στην 171 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 175. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 172 και 173. Αυτές οι δύο είναι ταυτόσιμες. Ονομαστική ψηφοφορία από τους πρασίνους. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε για την 181 άρχιδη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 Έχει αποσυρθεί 184, όχι 183, την ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είχε αποσυρθεί λοιπόν η 184 που ήταν ταυτόσημη, 8 του συγητή υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 185 υπέρ. Μάλλον καταπίπτει, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 με προφορική τροπολογία παριθμών 8 του κυρίου Ρικέ. Υπάρχουν αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία. Αν όχι, τότε ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 192 υπέρ, έχει αποσυρθεί 192 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 195 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 194 του κυρίου Τρεμόζα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 194. Νομίζω ότι εγκρίνεται άρτη ψηφοφορία για την 194. Πέρας. Όντως εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι επόμενες δύο καταπίπτουν, επομένως περνάμε στην 200 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε για την τροπολογία 12 του εισηγητή, 11 με συγχωρείτε του εισηγητή άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν εγκαταλείψει Μάικλ, εκτός από τους σκιώδης βλέπω. Εγκρίνεται πάντως. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 καταπίπτει, γιατί εγκρίναμε την 11 λέει ο πρόεδρο. Άρα περνάμε στην τροπολογία 204, όχι καταπίπτει και αυτή. Όχι, 204, τον κύριο Γκρός. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 205, η 206 και η 207 είναι ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 12 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές, ας ελέγξουμε για την τροπολογία 12 του εισηγητή άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 209. Ελέγχουμε τη 208 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 209 του κυρίου Κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την τροπολογία 209 παρακαλώ. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 212 του κυρίου Ζήλε υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 212 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 213 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 και η 13 καταπίπτει, η 214 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 217 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 218 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 219 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 220 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για την 221 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 223 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 227 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 239. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 240 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε για τη 240 άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένας επιπλέον ψήφος από το ΕΛΚ. Ματιέ. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά, εγκρίνεται. 241 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 242 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 244 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 246 καταπίπτει, η 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 247 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 249 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε για την τροπολογία 249. Μόνο ο κύριος Τρεμόζα ψήφισε. Άρτη ψηφοφορία για τη 249. Πέρας. Εγκρίνεται. Κύριε Τρεμόζα είχατε δίκιο, δεν είχαν ψηφίσει όμως όλοι. Τροπολογία 250 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, νομοθετική πρόταση υπέρ, άρτη μάλλον συγγνώμη, άρτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 36 υπέρ, 6 ψηφί κατά, μία αποχή εγκρίνεται λοιπόν νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 36 ψήφοι πέρ, 5 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας, την κυρία Σερακιάνη. Μην εξαφανιστείτε, αγαπητοί φίλοι, γιατί έχουμε και άλλες ψηφοφορίες. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Έχει κλείσει το μικροφωνό το πρόεδρος, δεν τον ακούμε. Ωραία. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, υπήρξε κάποια σύγχυση για την προφορική τροπολογία των πρασίνων, προκειμένου να προσθέσουμε τη λέξη rescue, σωτηρία. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια προσθήκη στη συμβαστική 1, ώστε να μην ε, υπάρξει κανένα πρόβλημα με, την, ε, με τον κατάλογο ψηφοφορία που, που μοιράστηκε χτες. Οι πράσινοι λοιπόν προσθέτουν τη λέξη rescue, την οποία προσθέτουμε στη συμβαστική αριθμό 1. Τροπολογία 72 έχει αποσυρθεί, οπότε πάμε στη συμβαστική αριθμό 1 κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, «οποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροποποίηση, σας ε, είπα του κυρίου Τέιλορ, με το rescue, rescue end, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Ωραία. Η προφορική τροπολογία λοιπόν περνά στην ψηφοφορία τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8. Καταπίπτει. Τροπολογία 74 επίσης καταπίπτει. Πού φτάνουμε τώρα. Η 11 επίσης καταπίπτει. 76 τώρα, στο άρθρο 1. Υπέρ παρακαλώ του κυρίου Τέιλορ. Ε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ένβι 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένβη 10. Καταπίπτει. Η τροπολογία 79 τώρα. Α, καταπίπτει και αυτή. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική αριθμός 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ενενήντα είναι η επόμενη. Με προφορική τροποποίηση του ΕΛΚ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία ε, α. Δεν υπάρχει αντίρρηση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ για την 92. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 93 καταπίπτει. NV11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 με προφορική τροποποίηση του ΑΛΔΕ. για να πάει στο άρθρο 2 παράγραφος 4β αν ψηφίσετε ναι ε, λέτε να μπει σε κάποιο άλλο σημείο αργότερα αν δεχτείτε την προφορική ε, τροπολογία είναι για να μπει αργότερα, έτσι. Δέχεστε την προφορική τροπολογία πρώτα απ' όλα, ναι. Ωραία, για αργότερα. Εντάξει, αργότερα λοιπόν. 97, Bilbao. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 κατά πίπτη, 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε παρακαλώ για τη συμβαστική 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Οπότε... Εκατόν δύο. Έτσι δεν είναι. Τι ψηφίζουμε τώρα. 104 είναι η επόμενη. Τέιλορ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενβι, 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το περίφημο πρόβλημα του safety και security, ποιο είναι ασφάλεια, ποιο είναι προστασία. Ψηφίζουμε τώρα όλη την τροπολογία, μια που συμβαστική απορρίφθηκε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ο κατάλογος ψηφοφορίας των σοσιαλιστών δεν είναι έτσι όπως πρέπει. Όπως αυτά που ψηφίζουν. Να μου δώσετε το δικό σας. Α, καλά, εντάξει. Να πάρω του ΕΚ τότε. Ναι. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 με κατατμήματα, πρώτο τμήμα από τους σοσιαλιστές, δραστηριότητα της υπηρεσίας. Το πρώτο τμήμα είναι αυτό. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της υποφορίας. Εγκρίνεται. Το υπόλοιπο του κειμένου τώρα υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 με προφορική τροποποίηση συγκητή και της Άλλη ιπέρ. Κατά από χέρε ενγκρίνεται. 114 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 τώρα, υπέρ, κατά, να ελέγξουμε παρακαλώ γιατί είναι 114. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία Β κατά τμήματα από το ECR. Πρώτο τμήμα το κείμενο χωρίς αυτό που λέει αξιολογώντας ε, τα κράτη-μέλη κλπ. Λοιπόν, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα δεύτερο τμήμα με τις λέξεις αυτές υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία γάμα Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένβη 13. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ε, όχι. Κατά πίπτη μου λένε. 119 τότε κατά δύο τμήματα. Εκτός από τη λέξη national, εθνικό, και μετά με τη λέξη. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 122 κατά τμήματα. Πρώτη ψηφοφορία είναι η λέξη May. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, όταν αυτό ισχύει, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ο κύριου Τέιλορ τώρα, 123 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Χωρίς τη λέξη solely. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ενβι 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 15 NB υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 NB υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 127 και 128 καταπίπτουν, οπότε ερχόμαστε στην 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 131 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Referred στο άρθρο 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένδυ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ για την 132 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 20 παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίπτεται. 134. De Grandes υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμόν 6. Δύο τμήματα. Υπέρ, δεύτερο τμήμα μάλλον, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 137 παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμών 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Του εισηγητή 23 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 8 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. προπολογισμό 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Προπολογισμό 8 τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία D, δέλτα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την προφορική τροπολογία δέλτα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις προφορίες. Απορρίφθηκε. 139 υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 139. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε για την 27 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε για την 18. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 140 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προπολογισμών 11 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 141 υπέρ. Η εγκρίθηκε όμως. 141 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 28. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 19. Από την NV. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία NV19. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη φοφορίες. Απορρίφθηκε. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προπολογισμών 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 προπολογισμών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προϋπολογισμό 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 προπολογισμών. Πρώτη πρόταση όμως καταπίπτει. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μα πόσες σελίδες έχουμε ακόμα, λέει ο πρόεδρος. Και ξεφυσάει. Τροπολογία 29. Υπέρ. Ναι, πάντα Ακόμα στο άρθρο 1 είμαστε. Ναι, 29 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 29. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 30. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προϋπολογισμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 ένβη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένβι 2 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 53. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι πέραστη της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τρία. Τη συγκητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε και την 56 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 4 καταπίπτει. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV3. Καταπίπτει. 5 επίσης. NV4 επίσης. Οπότε φτάνουμε στην 58. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Εισήγητη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Εισήγητη υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την τροπολογία 7. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 21-21. Τροπολογία 8 κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτα υπέρ, πρώτο, πρώτο υπέρ, κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 21-21. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται, ναι. Οπότε καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61. Κατά τμήματα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 62 καταπίπτει. 60 τώρα με προφορική τροποποίηση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει, σωστά. Envy 5 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9. Α, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 68. Ωραία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντεύουμε. Κοντεύουμε. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. προϋπολογισμών 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα τώρα, ένα α νέο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροποποιημένη πρόταση λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρα τη ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 5 κατά και 2 αποχές. Εγκρίθηκε και το νομοθετικό ψήφισμα. Τώρα ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν και συγχαρητήρια στον εισηγητή. We have One, two, three. Πάμε τώρα στην ε, χμ, λέει ο πρόεδρος. Okay. So we still got some more votes to... Έχουμε κάτι ακόμα ψηφοφορίες να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τραβάμε κουπί. Εδώ έχω την, δεν ξέρω αν είναι σωστή σειρά, έχω την Γεωργία. Μία ψηφοφορία μονάχα, ο κύριος Σούλ ο εισηγητής. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για το σχέδιο έκθεση για την κοινή αεροπορική συμφωνία με τη Γεωργία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψήφισατε όλοι. Όλοι. Όλες. Πέρα. Πέρας. Η Γεωργία θα χαρεί πάρα πολύ, διότι πέρασε με 38-2 αυτή η, η έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Ούλμερ. Ευρωμεσογειακή Συμφωνία με το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας. Άρχεται η ψηφοφορία, η κυρία Σένα Λόβα είναι η συγκέντρια. Άρχεται η ψηφοφορια ψηφιζα Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 37-1. Ευχαριστώ την κυρία Λόβα. Η έκθεσή μου τώρα για την Σύμβαση των Αθηνών σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά πιβατών και των αποσκευών τους. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 39. 0. Μία αποχή. Θα βρω ποιος το έκανε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην έκθεση, στη γνωμοδότηση μάλλον του κυρίου Μαρινέσκου για την πολιτική ανταγωνισμού. Τροπολογία 1, τεμπάκερ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος βεβαίως ε, βεβαίως ελέγχουμε την τροπολογία τέσσερα. αρχή την ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται Συμβαστική τροπολογία την 5, 6, 7, 8 αλλά και 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Πάμε στη 10. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 12 έχει εκπέσει. 13 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 σε δύο τμήματα πρώτο κομμάτι διαγραφή ενός, ε, ενός τμήματος Το δεύτερο υποστηρίζει την αγορά. Λοιπόν, ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματο Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Μια διευκρίνηση στον κατάλογο ψηφοφορίας λέει ότι καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία η οποία έχει εγκριθεί. Νομίζω ότι και αυτό το εγκρίναμε. Είμαστε συνεπείς λοιπόν. Όχι, όχι. Είναι πρόσθετο η διαγραφή ενεκρίθη. Είναι συμβατή με την συμβαστική τροπολογία, αλλά <clears throat> μπορούν να συμβαδίσουν και τα δύο. Κύριε Μαρινέσκου, το κείμενο από το δεύτερο τμήμα είναι ταυτόσιμο με το κείμενο από τη συμβαστική τροπολογία, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Ίσως δεν έπρεπε να ψηφίσουμε γιατί το είχαμε ψηφίσει, αλλά τώρα είναι σαφέστερα τα πράγματα. Ωραία. 16 Γιατί δεν εκρίθη όλοι 15. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. 16. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 16. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Μπαχ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε τη 19 παρακαλώ γιατί κανείς δεν σηκώνει το χέρι του πια άρχεται για τη 19 ως προστίκη πέρας εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 με προφορική τροποποίηση από τον εισηγητή. Με την προφορική τροποποίηση ψηφίπερ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές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 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας 35-3 εγκρίνεται. Με δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μαρινέσκου. σχέδιο γνωμοδότησης για μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγητής είναι ο κύριος Ζασάρα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τέσσερα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Έξι. χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Εφτά. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 προφορική, προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 1 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 18 με την προφορική τροποποίηση ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 20 εκπίπτει και την 18 τελευταία ψηφοφορία Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται 37-2 χωρίς αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ζασάδα. Ως εκ τούτου. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε τον κύριο Ζεμπόφσκι στις 3 η ώρα, το συντονιστή της ΦΑΠ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως όλους σας και όλους τους εισηγητές για τη συνεργασία σας σήμερα το πρωί, γιατί καταφέραμε να κάνουμε μια δύσκολη και μακρά ψηφοφορία. Ευχαριστώ και τη γραμματεία, γιατί ήταν δύσκολη η ιστορία του ξεμπερδέματος των τροπολογιών. Τα καταφέραμε, αλλά σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Καλό μεσημέρι.